Buenas tardes. Buenas tardes, silencio por favor. Γεια σας, γεια σας λοιπόν, καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ. Se reanuda συνεχίζουμε την συνεδρίαση. Απλώς υπάρχει ένα θεματάκι πριν συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Γιατί η γραμματεία μας που είναι τόσο αποτελεσματική μου υπέδειξαν ότι κάναμε ένα λάθος κατά την ψηφοφορία. Αφορά... Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα άλλο, πρέπει να το ξέρετε. Πρόκειται τη συμβαστική υπαριθμών 32 στο τμήμα υπαριθμών 8 είχαμε προφορική τροπολογία και είχε υποβληθεί ένσταση κατά τη ε, ψηφοφορία με την προφορική. Και όμω, ε, από δικό μου λάθο, την ψηφίσαμε. Οπότε, ε, επομένω, το, το, αυτό το κομμάτι όσο περιέχεται στο, 7 και άρα το, το, 8 θα θεωρηθεί ότι δεν ψηφίστη παρά το, αντίθετο. Το 8, το τμήμα 8 της συμβαστικής 32 ως μη γενόμενο. Και Οπότε τώρα είσαστε εδώ για να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα. Θα ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση ως τροποποιήθηκε. Και άρχεται η ψηφοφορία. Bueno, no cerramos, comienza. Vale. Ναι, τώρα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Έχουμε μία ψήφο σοσιαλιστική επιπλέον. πάμε πάλι. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Θα το ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Δύο τώρα λέει. Εκτός μικροφώνου. Για να επαναλάβω την ψηφοφορία.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 15 κατά 9 και μία αποχή εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα ε, από την ε, τους ε, επιτροπή των προπολογισμών υπαριθμών 1 ψηφίζουμε πέρας Απροβάδα. Εγκρίνεται. Budget 2. Προπολογισμοί 2. Comienza. Cerramos. PP tiene uno de más. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Απροβάδα. Εγκρίνεται. No. Ρέτζι, υπαριθμόν 1. Ψηφίζουμε. Bien. Termina. Rechazada. Απορρίπτεται. Και εν τέλει θα ψηφίσουμε την ε, νομοθετική πρόταση εις το σύνολό της. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι.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 Si hay 14, 10 y 2 son 26. Θα τις κάνουμε και πάμε 14, 10 και δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Είμαστε 15, βγήκαν 26. Πάει ένας παραπάνω από την ενωτική αριστερά. Θα την ξανακάνουμε. Llevamos, hemos votado mil veces hoy. En la última vamos a ver si cada uno vota lo que tiene que votar. Ε, αλλά τόσες, τόσες, τόσες χιλιάδες σήμερα δεν πειράζει. Ας κάνουμε σωστά την... Ε, έγινε και ένα λάθος στο τέλος. λέει ένα λάθος έγινε, αλλά είναι από την ΚΟΕ. Τέλος πάντων, ψηφίζουμε τώρα. Cierra. Ahora, 13 votos a favor, 10 en contra. 13-12. Εγκρίνεται. Bueno, una vez finalizado, a mí sí me gustaría, un momento de silencio por favor, darle por supuesto la enhorabuena a la ponente, como siempre se hace cuando se... Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και βέβαια συγχαρητήρια σε όλους εσάς για το πώς έχουμε διεξαγάγει την ψηφοφορία και για το Μπράβο σε που μας βοήθησαν για να μπορέσουμε να κλείσουμε τους συμβασμού, να κάνουμε τι εφορίε αυτέ. και φυσικά και το επιτελείο μα εδώ από τη Γραμματεία, γιατί χωρί τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου. Y recuerdo que la comisión sigue.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 combination of that. So. Por favor. Quiet, please. Por favor. Por favor, la comisión sigue. Συνεχίζουμε τη συνεδρία τη Επιτροπή.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 Μια στρατηγική για την Αγγλία συνεδριτεί και το Ιωνικό Πέλαγος. Η συγκεκριτή είναι ο κύριος Μιλάνα, ο αντιπρόεδρος Μιλάνα. Un primer intercambio de opiniones con una breve presentación por la Comisión Europea de la Comunicación. Έχουμε επομένω, εκτό από την εισήγηση του εισηγητού, έχουμε και την ανακοίνωση τη 3η Δεκεμβρίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μιλάνα. κάνεις λοιπόν, για αυτή την παρουσίαση που είναι η πρώτη ευκαιρία την οποία τη συζητούμε όσον αφορά αυτό το σχέδιο έκθεση. Και κατά τον τρόπο να τα πούμε αργότερα, για να δούμε το περί τίνο πρόκειται. Πρόκειται για το πώ θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία. Για συμπαθάτε με λέει ο να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία και στην οποία και να εντάξουμε είναι κάτι το οποίο έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από πολλέ οπτικέ γωνίε, μια στρατηγική που να καλύπτει την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγο για αυτή την περιοχή. Και επίση ακριβώ πρόκειται για την αλία που έχει δύο σε αυτή την περιοχή. Διότι εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικές προβληματικές. Πρώτα πρώτα υπάρχει σε αυτή την περιοχή μια συνύπαρξη ε, των κοινοτικών και των μη κοινοτικών χωρών και κάποιες ε, χώρες οι οποίες είναι καθοδόν για την ένταξη. Δεύτερον, ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτές τις θάλασσες ας πούμε, έχουν είναι ριχά τα ύδατα, επίσης έχουμε γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι τελείως διαφορετικά ε, από την υπόλοιπη Μεσόγειο, όμως ε, ισχύει το ίδιο καθεστώς, τους ίδιε κανόνε κανόνες εκεί όπως και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να καταρθεί μια προσπάθεια να μπορέσουμε να χαράξουμε μια στρατηγική η οποία κατά κάποιο τρόπο να καταστήσει αυτή την περιοχή ως περιοχή πιλωτική όπου να είναι δυνατόν να θεσπιστεί μια στρατηγική, μια πολιτική τέτοιου είδους και να έχουμε εδώ πέρα συντήρηση, διάσωση λευτικών πόρων μια που σοβεί αυτή η κρίση και πολύ σοβαρή στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει, με το ερώτημα που θα καταβάλουμε τους αμέσως σε επόμενες εβδομάδες και μήνες, να έχουμε τι θα, να δούμε τι θα κάνουμε με την υπάρχουσα νομοθεσία και να δούμε πώς θα εντάξουμε σε αυτές τις ε, στρατηγικές, την ολοκληρωμένη στρατηγική, με αυτές τις επιλογές που τώρα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής δηλαδή. Και ζήτησα να γίνει αυτή η έκθεση γιατί έχουμε κρίση στην αλία της Μεσογείου και αυτό έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη κρίση της αλίας Βεβαίω όμως σε αυτή την περιοχή υπάρχουν ιδιαίτερε δυσκολίες από πλευράς ε, ε, αλληλευτικού κλάδου και επομένως ε, πρέπει με κάποιο είδους παρέμβαση στα όσα τώρα προβλέπονται να δούμε πώς θα έχουμε ε, καλύτερη απόδοση, καλύτερο εισόδημα και ε, παρέμβαση που θα βελτιώσει τους, την ε, συντήρηση των ελευθερικών πόρων. Οπότε, η εξατομίκευση, ας πούμε, κάποιων σημείων επί των οποίων θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί, αυτό ε, να μην θεωρηθεί ότι είναι εύκολο, τώρα θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά και επίσης έχουμε αυτή την ε, δύσκολη προβληματική για αυτές τις περιοχές το, το, το, το ότι δηλαδή αυτές οι περιοχές της ε, Μεσογείου είναι όμορες με κάποιες άλλες γιατί, γιατί έχουμε στην Μεσόγειο 8 κοινοτικέ χώρες αλλά έχουμε και άλλες 14 που δεν είναι μέλη κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε οποιαδήποτε πολιτική ας το πούμε λιτότητος και οποιαδήποτε αυστηρία στην πούμε, πολιτική ε, δεν πρέπει να προσκρούει στο τι ισχύει στην περιοχή αυτή οπότε ακριβώς πρόκειται για μια περιοχή με τις δικές της ιδιομορφίες επίσης η Αδριατική είναι ο χώρος όπου εκεί πέρα κάνουμε κάποιο είδους πειραματισμό για αυτές τις νέες σχέσεις γιατί έχουμε εκεί πέρα κοινωτικές και μη κοινωτικές χώρες που βρέχονται από αυτή την Αδριατική που δεν είναι και πολύ μεγάλη οπότε εκεί μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιο είδους διεθνείς συμφωνίες για την Αλία και ε, πρόκειται ουσιαστικά για απόπειρα διαχείριση κάποιων ελευθερών πόρων που ανήκουν σε κάποια άλλη χώρα. Και επίση έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τι ε, προποθέσει, ούτω ώστε να μπορέσουμε με αυτές, τι τις να, να συμβάλλουν και να έχουμε μία θετική συμβολή στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουμε δηλαδή επίσης θετικό αντίκτυπο με τα μέτρα μας αυτά στους αλληλευτικούς πόρους. Άλλο στοιχείο τώρα που πρόκειψε αυτή την αξιολόγηση είναι το τι περί τι είδους θάλασσα πρόκειται, ποια, ποια θάλασσα προσφέρεται για τέτοιου είδους προγραμματισμό. Βέβαια και αυτό το επιχείρημα καλύπτεται από κάποια πρόσφατα έγγραφα Κοινοβουλίου, Επιτροπής και αφορά αυτή την ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική μεταβλητή. Οπότε και αυτόν τον τρόπο τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε όσο είναι καλύτερα τη θάλασσα και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που επιδέχονται η αλία, που όχι, που θα γίνεται η δατοκαλλιέργεια που τουριστικές δραστηριότητε που θα πρέπει να υπάρχουν οι βασικοί κόμβοι των μεταφορών που θα μπορεί να ασκεί την ενεργειακή πολιτική οπότε θα πρέπει να συμπληρώσουν προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τελικά να επιλεγεί μια πρόταση την οποία θα εξετάσει τη δομήρηση του Κοινοβούλιο. Και προβλέπεται πρικοδότηση ικανή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο πιο δοκιμό τρόπο, ώστε αυτέ οι δραστηριότητε να έχουν βιώσιμο χαρακτήρα και θα, να είναι ε, εφαρμόσουμε τόσο προβλέπονται. Οι δε υδατοκαλλιέργειε, να δούμε κατά πόσο γίνεται να αναπτυχθούν σε τρίτα κράτη. Και οπότε να δούμε όλε τι συνθήκε με τι οποίε θα ισχύσουν οι, οι κοινοτικέ και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με αυτές τις τρίτες χώρες οπότε όλα αυτά να οδηγούν σε επενδύσεις στην Ευρώπη παράγουμε 1 εκατομμυριο κοκκί κοκκινικόμε 25-250.000 τόνους ε, ηχθείων και καταναλώνουμε 5 εκατομμύρια τόνους. Άρα, εισάγουμε con l'assenza eh, di regole, spesso con eh, problemi che più volte abbiamo affrontato. Εισάγουμε το υπόλοιπο, επομένω. Γι' αυτό έχουμε προβλήματα οποία επανειλημμένω, τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων από αυτόν. Και ελπίζω αυτά που θα πείτε θα συμπληρώσουν το έργο μου. Και με διαδικέ ε, συναντήσεις όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να, να, να φτάσουμε στο αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν και μετά στους υπόλοιπους βουλευτές που θέλουν να λάβουν το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ενάδεια. Bueno, pues sorprendentemente, sí. Ευχαριστώ πολύ. Στις 3 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και βασίστηκε ε, στις συζητήσεις που έχει με τους φορείς της Αδριατική και του Ιωνίου Πελάγους, όπως επίσης και των ενδιαφερόμενων στα, που συμμετείχαν στα τρία σεμινάρια που κάναμε το 2012 στην Αθήνα, στην ε, Τεριέστη και στο Πορτορούς. Η ανακοίνωση αυτή είναι μια αφετηρία. Μετά θα περάσουμε στο σχέδιο δράσης θα ορίσουμε το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες του χρόνου. Και όπως ξέρετε και εσείς, το σχέδιο δράσης είναι ένα κυλιόμενο έγγραφο το οποίο συνεχώς ενημερώνεται. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιουνίου. Στην ανακοίνωση δηλώνεται απερίφραστα πως εάν τα κράτη-μέλη ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει στρατηγική για την περιοχή αυτή, τότε η θαλάσσια αυτή στρατηγική θα αποτελεί και το πρώτο σκέλος ε, αυτού. Η στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Είναι η μπλε ανάπτυξη, ε, το υγιές ε, ε, θαλάσσιο περιβάλλον, οι πιο ασφαλείς θάλασσες, και οι βιώσιμες και η βιώσιμη και υπεύθυνη αλληλεία. Οι τέσσερις αυτοί οι πυλώνες θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες προτεραιότητες με τις σχετικές δράσεις και με τα εμβληματικά πιλωτικά ε, προγράμματα τα οποία θα μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα χρηματοδότησης ε, για τις περιφερειακές αυτές στρατηγικές αλλά και από το Horizon 2020. Αυτές είναι κάποιες από τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Άλλες ενδεχόμενες πηγές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι διεθνείς φορεί, για παράδειγμα το ε, επενδυτικό πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως επίσης και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Τώρα που επιλέξαμε τους χώρους στους οποίους θα συνεργαστούμε, περιμένουμε τις ιδέες για τα συγκεκριμένα project, τα οποία έχουν αρχίσει και καταφθάνουν. Οι προτεραιότητε μα αποτελούν το απόσταγμα αυτών των προτάσεων και θα έχουμε, επαναλαμβάνω, και κάποια που θα είναι εμβληματικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η στόχευση, χωρί να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με μια. για τα όσα είπε ο κύριος Μιλάνα, να σας πω πως τον πυλώνα για την πλέον ανάπτυξη η υδατοκαλλιέργεια θεωρείται ως ένας από τους κλάδους με το μεγαλύτερο δυναμικό για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιουνίου. Η υδατοκαλλιέργεια είναι ο κλάδος, ο διατροφικός κλάδος, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αλλά αντίθετα με τις παγκόσμιες τάσεις, η ευρωπαϊκή παραγωγή βρίσκεται σε τέλμα. Και αυτό βεβαίως επειδή αντιμετωπίζονται και κάποιοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί κοινοί για όλες τις χώρες της Αδριατικής και του Ιωνίου. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με το σχεδιασμό για τη βιωσιμότητα και να επιτρέψουμε να ε, ε, ε, επεκταθεί η υδατοκαλλιέργεια είτε σε μακρινές απομακρυσμένες περιοχές είτε σε απομονωμένες περιοχές όπου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μικρότερες. Και εδώ χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Μπορούμε να το δούμε και με το θέμα της θαλάσσιας χωροθέτησης και χωροταξίας. Για την αλληλεία, οι προτάσεις μας και τα όσα προτείνουμε με την αναθεώρηση είναι γνωστά. Προσθέμενη αξία στα προϊόντα αλληλείας και κυρίως από την μικρή κλίμακα αλληλεία, ε, συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, τις τοπικές ομάδες δράσης και τους αλληλείς, ε, πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών οργανισμών και ε, αλληλευτικών εταιριών. Δράσεις που θα μπορούσαν να εκπονηθούν στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής θα μπορούσαν στρατηγική στρατηγικής, στρατηγικές εμπορικής ανάπτυξης ε, που να προτιμώνται και να προκρίνονται τα τοπικά ε, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τα ΛΟΔΑΠΑ, οργάνωση τοπικών εκθέσεων ε, και βεβαίως ανάπτυξη νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον λόγοι για τους οποίους το Ιόνιο και η Αδρετική θα δρέψουν τα πλεονεκτήματα μιας τέτοια στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή θα μας επέτρεπε να βρούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για την ανάπτυξη και την απασχόληση που συγκεκριμένα αναφέρονται σε αυτές τις δύο θάλασσες. Στις 8 Οκτωβρίου στην Κύπρο ε, υιοθέτησαν τα κράτη-μέλη την σχετική ατζέντα στα πλαίσια της ε, για το 2020 με την δήλωση της ε, Λεμεσού, έτσι ώστε ο κλάδος να ενισχυθεί, όπως θα ενισχυθούν και ο τουρισμός παράλληλα και οι μεταφορές. Η λιγότερο εκμεταλλευ... οι κλάδοι που βρίσκονται υπό μικρότερη εκμετάλλευση σήμερα ενδεχομένως να πρημοδοτηθούν έτσι ώστε να έχουμε κάποιες τεχνικές καινοτόμες δατοκαλλιέργειες παράλληλα με τις ΑΠΕ και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Χρειαζόμαστε λοιπόν περιφερειακή συνεργασία για να λάβουμε υπόψη τις ιδιάζοντες ανάγκες του τοπικού πληθυσμού που θα βρεθούν πια στο κέντρο των ε, προτεραιοτήτων μας. Χρειαζόμαστε συνέργεια και βέβαια ε, να λαμβάνουμε υπόψη και να συνεργαστούμε συμμορφωνόμαστε με την επικουρικότητα. Η θαλάσσια στρατηγική θα φέρει πλεονεκτήματα και η μακροπεριφερειακή στρατηγική θα εξασφαλίσει τη σύνδεση μεταξύ κλάδων και δραστηριοτήτων, αρκεί όλα τα προγράμματα να ευθυγραμμίζονται και να ακολουθούμε και ακόμα εγκάρσια σε όλες μας τις πολιτικές τους είδους κανόνες. Και αυτό πάντα διασυνοριακά. Τώρα, συγκεκριμένα για την αλληλεία, η ανακοίνωση για τις πρωτοβουλίες για την Αδριατική και το Ιόνιο θέτει τις εξής προτεραιότητες. Καταρχήν, βιώσιμη διαχείριση της αλληλείας και των αλληλευμάτων, πολυετή προγράμματα και μέτρα όπως οι προστατευόμενες περιοχές με την ευρύτερη έννοια συνεισφορά στην κερδοφορία και βιωσιμότητα της αλίας μέσω της ενίσχυσης, την εσπλοκή των ενδιαφερομένων στην διαχείριση της αλίας, έτσι ώστε να έχουμε βιώσιμα αλιεύματα και μη ρηπογόνες αληφτικές ε, δραστηριότητες, καθαρά ψάρια να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στη μεταφορά γνώσεων και καλύτερο έλεγχο των αληφτικών δραστηριοτήτων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επιστημονική συνεργασία για την αλληλεία έτσι ώστε να αποκριθούμε καλύτερες ανάγκες του κλάδου αλληλείας και Αν αμφίβολα, η δημιουργία μιας τέτοιας στρατηγικής εκ του μηδενός είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καθήκον και με ιδιαίτερη εκτίμηση αποτιμούμε το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Κοινοβούλιο εδώ όπως έγινε και για την περιοχή του Ατλαντικού. Αναμένουμε λοιπόν με προσδοκία τις προτάσεις τις οποίες εσείς θα μας υποβάλλετε για να στηρίξουμε τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφέρουμενους φορείς καθόλου αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέτσνερ είναι η πρώτη βουλευτής που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά τις ενοποιημένες πολιτικές, ε, αναγνωρίζω όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν, δεν είμαι πολύ καιρό εδώ, αλλά υπήρξα εισηγήτρια σε θέματα μεταφορών που είναι συνδεμένα. Νομίζω όμως ότι και αυτό το θέμα συνδέεται με την ενοποιημένη ναυτιλιακή πολιτική, την ενοποιημένη προσέγγιση. Διότι πιστεύω ότι η Ελία αποτελεί μέρος αυτής της ενοποιημένης ναυτιλιακής πολιτικής. Και αν στο μέλλον διαχειριστούμε και αναπτύξουμε με βιώσιμο τρόπο τις θάλασσες, πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς, ε, επειδή ε, η περιοχή αυτή ε, θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και όπως είπατε κύριε Σιγητά, ο τομέας του τουρισμού των ακτών, ο τομέας της κουραζιέρας, αλλά επίσης και αλίας και offshore αλίας. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους και τους θυγόμενους. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα και πρέπει να διαχειριζόμαστε τους πόρους με τρόπο αηφόρο βιώσιμο και να αλλιεύουμε μόνον ε, τις ποσότητες που θα επιτρέψουν να υπάρξουν ε, ψάρια για τις επόμενες Είναι Συνεπώς, ε, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Συχνά στη Μεσόγειο, οι ευθύνε και τα όρια δεν είναι τόσο σαφή. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ποιο θα διαχειρίζεται ποιον τομέα, είτε πρόκειται για την αλία, είτε για την υδατοκαλλιέργεια. Για την υδατοκαλλιέργεια συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζουμε ποιο θα εκμεταλλεύεται τι. Δεν πρέπει να τα αναμειγνύουμε μεταξύ του αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως. Μερικέ φορές πρέπει να δούμε και τα ολικά πάρκα offshore, πώς θα έχουν τοποθετηθεί, ώστε να μην βλάπτουν την αλεία. Ε, πρέπει να εξασφαλίζουμε και μια οικονομική βιωσιότητα. Η η δαδικαλλιέργεια είναι απαραίτητη για την μπλε ανάπτυξη. Σε άλλες περιοχές του κόσμου, το 50% ε, των ψαριών που κατανάλλονται προέρχονται από την εδωκαλλιέργεια, ενώ εμείς έχουμε χαμηλότερο ποσοστό. Συνεπώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη εδώ. Ε, όλα τα θέματα που σχέση με τη θάλασσα και την ελία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αλλά δεν θα μακρηγορήσω. Θα γράψω κάτι όμως, ναι αλλά όχι πριν από τα Χριστούγεννα, για του χρόνου. Ναι, θα συμμετάσχω με μεγάλη χαρά σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φράγα. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση να κάνω. Μιλάμε για θαλάσσια στρατηγική, για το Ιόνιο και την Αδριατική, αλλά στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο αυτό, έτσι νομίζω ότι έτσι, πώς διαβάζω εγώ το κείμενο, λέει αλλιευτική στρατηγική και όχι θαλάσσια στρατηγική. Δηλαδή, θα μιλήσουμε μόνο για την αλληλεία ή μιλάμε για κάτι πιο ευρύ, δηλαδή κάτι διαφορετικό, γιατί εσείς μιλάτε ε, για θαλάσσια στρατηγική και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ανακοίνωσή της. Αλλά εδώ στην ημερησία διάταξη λέμε αλλιευτική πολιτική ε, για την ε, περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν ε, ξεκαθαρίσαμε τι συμβαίνει, διαφορετικά δεν καταλαβαίνω γιατί ακριβώ μιλάμε. Στρατηγική για την αλληλεία, λέει η Μερίσια Διάταξη. Νομίζω πω ο εισηγητή είναι ο πιο κατάλληλο για να το απαντήσει. Ο κύριο Μιλένα. Θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θέλετε, ή σε όλα τα άλλα ερωτήματα. Κύριε Μιλάνα. Τέλος, να γίνω ερωτήματα, δεν απαντήσω σε αυτό. Κύριε Μιλάνα, τι είπε η κυρία Φράγα, το ακούσατε. Μπορείτε να τις απαντήσετε. Αλλιώς θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα απαντήσει κάποιος άλλος. Και θα σας δώσουμε το λόγο κλείνοντας. Άρα λοιπόν μάλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιστρέψω το λόγο. Well, thank you very much. No, our communication... πολύ. Η ανακοίνωσή μας αναφέρεται ...την αλληλευτική στρατηγική. Περιλαμβάνει όμως ένα μεγάλο μέρος, το οποίο, όπως είπα, αφορά την αλία γενικά. Αλληλευτικά προβλήματα και αυτό είναι ένας από τους πυλώνες από ό,τι καταλαβαίνω. Συνεπώς θα αποτελέσει μέρος αυτής της ευρύτερης ναυτιλιακής στρατηγικής. Ως προς την αλία γενικά, υπάρχει, το έργο το οποίο επιτελείται στα πλαίσια της Επιτροπής Αλίας στη, Μεσόγειο, όπου προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη διαχείριση πόρων σε περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριμένα σχεδιάζουμε φέτος να προτείνουμε Ε, τη μελέτη της δημιουργίας μακροχρόνιων σχεδίων ανάπτυξης στην Αδριατή και, αλλού για τα μικρά πελαγικά είδη. αυτό είναι ένα από τα είδη που είναι σημαντικά ε, ψάρια για την Ιόνιο και την Αδριατική. Επίσης, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που προβλέπει ο Μεσογειακός Κανονισμός για να προτείνουμε μακροχρόνια ευρωπαϊκά σχέδια διαχείρισης αυτό προβλέπεται ήδη από τους μεσογειακούς κανονισμούς και είναι ένας τομέας όπου υπάρχει περιθώριο για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκού προγράμματος, κυρίως για τα μικρά πελαγικά είδη ε, στην ε, Αδριατική και τον Ιόνιο Πέλαγος. Πολλά έρχονται στο νου μας, πολλά μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε σε αυτά τα πλαίσια. Όπως γνωρίζετε και είπα πρωτήτερα, μια τέτοια στρατηγική κατά κάποιον τρόπο ε, είναι μια στρατηγική την οποία ξεκινάμε εμείς και αν θέλετε θέλουμε να ζητήσουμε στα κράτη-μέλη και στους ενδιαφερόμενους να κάνουν προτάσεις, να παρουσιάσουν προγράμματα και είμαστε διατεθειμένοι να τα υποστηρίξουμε. Γι' αυτό μπορείτε εσύ να μας βοηθήσετε για να τονώσουμε αυτή τη συζήτηση σε τοπικό επίπεδο με τους τοπικούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους ώστε να προτείνουν ιδέες με βάση, βάση των οποίων μπορούμε να ε, κινητοποιήσουμε και να συγκεντρώσουμε τα κεφάλαια που θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και ο κύριος Μιλάνα, τελευταίος ομιλητής, για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τη συζήτηση που έγινε και βέβαια στην... Εδώ υπάρχει ένα διφορούμενο. Έχουμε μια στρατηγική για την Αλία, στην Αδριατική και στο Ιόνιο Πέλαγος. Τι συνέβη αφού του ζητήσαμε αυτή τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή, χωρίς να το γνωρίζουμε, κατέθεσε μια στρατηγική για το Ιόνιο Πέλαγος και την Αδριατική και είναι αυτό το ε, για το οποίο μιλήσατε εσείς. Για το άλλο έγγραφο όμως, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή, νομίζω ότι θα έπρεπε εμείς ως Επιτροπή Αλίας να ζητήσουμε μία ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών, διότι ως ήθιστε ένα έγγραφο για την ενοποιημένη ναυτιλιακή πολιτική αφορά σε μεγάλο βαθμό και την Αλία. Συζητείται όμως μόνον στην Επιτροπή Μεταφορών, παρά το γεγονός ότι Προ δύο ετών είχαμε μια παρόμοια διαμάχη πάνω ε, σε ένα άλλο θέμα και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα από αυτού. Γι' αυτό παρακαλώ τους συντονιστές να φροντίσουν να ληφθούν τα σχετικά μέτρα, διότι μιλάμε για δύο ξεχωριστά έγγραφα. Καταλαβαίνω αυτό που μας είπε η Κομισιόν, αλλά ίσως μια άλλη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ε, θα παρουσιαστεί σε μια άλλη στιγμή της συζήτησης του κειμένου το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί αλλού στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν υπήρξα σαφής, αλλά για μας τουλάχιστον η έκθεσή μου θα είναι μια έκθεση για την αλληλευτική στρατηγική ε, στην Αδριατική και στο Ιόνιο Πέλαγος. Δεδομένου ότι δεν πρέπει να ε, στρουθοκαμιλίζουμε εάν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και άλλες μελέτες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα εδώ. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μεγάλος πυλώνας της Αλλά μιλάμε για ενδιαφερόμενους, για εμπλεκόμενους, για επιστημονική συνεργασία. Σε αυτό το έγγραφο όμως δεν γίνεται λόγος για τις σχέσεις με τις μη κοινωτικέ χώρες. Και αυτό προσπαθούσα να πω πρωτήτερα. Αποδίδω πολύ πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις χώρες για τη Μεσόγεια. Μπορούμε να έχουμε όση βιωσιμότητα θέλουμε από πλευρά Ιταλία, Σλοβενία, Αδριατικής. Αν όμω απέναντί μα έχουμε εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν καταστροφικά μέτρα, τότε και κατασκευάζουν ή μάλλον δημιουργούν έναν ανταγωνισμό χωρίς κανόνες, ε, διότι δεν τους αφορά αυτή η αγορά, η αγορά είναι δική μας, τότε τα πράγματα θα είναι σοβαρά. Και πιστεύω ότι δεν μπορούν να είναι απόντες αυτοί στις προτάσεις της Επιτροπής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τρίτες χώρες. Και πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν μπορεί οι τρίτες χώρες ε, να είναι μόνο μέρη σε διεθνείς συμβάσεις. Ναι. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα προβλέπονται στις συμβάσεις, αλλά αυτά δεν αφορούν τη στρατηγική η Μεσόγειος έχει ανάγκη μιας εξωτερικής πολιτικής αλίας, διότι μπορεί οι οκτώ χώρες να συμπεριφέρονται θαυμάσια, αλλά εάν δεν παρέμβουμε με πολύ πιο σημαντικές πολιτικές ενέργειες στη Μεσόγειο, ενέργειες που έχουν σχέση με τα αναπτυξιακά μας συστήματα. Στη Βόρεια Αφρική, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές αναπτυξιακές ενέργειες αλλά τα αναπτυξιακά μέτρα δεν έχουν σχέση με τους κανόνες μας. Θα τα ξαναδούμε αυτά. Επανέρχομαι τώρα στην έκθεσή μας. Περιμένω από όλους σας προτάσεις μετά από τα γεγονότα και θα ήθελα να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους και μετά τις γιορτές με τη νέα χρονιά θα δούμε με τους σκιώδεις συζητητές τι θα κάνουμε προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα σύντομο γραπτό κείμενο και να δούμε πώς τα πλαίσια αυτού του γενικού, του γενικού σχεδίου θα έχουμε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε η αλία να μην είναι η ευκαιρία να χρησιμοποιεί κανείς απλά και μόνο το Ιόνιο Πέλος και την Ενδρατική για να ψαρεύει, αλλά να έχουμε μια στρατηγική που ε, θα αναφέρεται ε, στην παραγωγή, στην ατοκαλλιέργεια, στην αλληλεία γενικά και στο σεβασμό των βιολογικών πόρων και ε, στη γενική βιωσιμότητα της θάλασσας, των δύο θαλασσών αυτών, υιοθετώντα ορισμένα κανονιστικά μέτρα που δεν υπάρχουν ακόμα και που είναι δύσκολο να διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ τη συμβολή σας. Αυτή η ανταλλαγή με την Κομισιόν υπήρξε πολύ χρήσιμη και ας αρχίσουμε τη δουλειά και αν έχετε προτάσεις θα τις ακούσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιλάνο. Θα περάσουμε λοιπόν στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού αριθμού 850 του 98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών. Σήμερα θα ακούσουμε την παρουσίαση που θα κάνει τις πρότασεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, μια έκθεση που θα αναλάβει ο κύριος Νικολέσκου, δεν το βλέπουμε εδώ ακόμα σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντωμεταξύ το λόγο. who is taking the floor from the Commission? Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σας παρουσιάσει μία πρόταση ε, που αποτελεί ένα κομμάτι της ε, εξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου, του screening. Προσπαθούμε λοιπόν να χωρίσουμε τις αρμοδιότητές μας σε κατεξουσιοδότηση ε, πράξης και μη. Και εφαρμοστικές λοιπόν είναι οι τροπολογίες στον κανονισμό 850 του 98 για την διατήρηση των ελευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών σύμφωνα με τους κανόνες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια καθαρή ευθυγράμμιση. Γι' αυτό και οι τροποποιήσεις που έχετε μπροστά σας δεν, οι τροπολογίες με συγχωρείτε, δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό αυτό και για τον κανονισμό 1435. Τι προτείνουμε λοιπόν με αυτή τη νέα πράξη. Προτείνουμε να κάνουμε μια νέα κατανομή των αρμοδιοτήτων που έχουν ε, ανατοθεί, ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμοστικές πράξεις και κατεξουσιοδότηση πράξης. Προτείνουμε λοιπόν για την κατανομή των περιοχών σε γεωγραφικές ε, περιοχές, για την τροπονοποίηση των ε, κανόνων ε, για την χρήση, και το συνδυασμό των θελασσινιδών, για τις τεχνικές περιγραφές και τη μεθοδολογία των εργαλείων που μπορούν να συναυθούν στα δίχτυα και τα ε, πια σκάφη τα οποία είναι μεγαλύτερο από 8 μέτρα στο μήκος μπορούν να φέρουν δοκότρατα ε, να είναι ε, κατεξουσιοδότηση πράξης όπως, κατεξουσιοδότηση πράξης, όπως επίσης την περίπτωση που έχουμε αλλαγές στη μεταναστευτική ροή των ηχθιδίων και οπότε αυτό επηρεάζει ε, της, ε, τη διατήρηση αυτών των πόρων. Για τις ε, εφαρμοστικές πράξεις προτείνουμε να έχει για κάτι τέτοιο η Κομισιόν στους τεχνικούς κανόνες που σχετίζονται με τη μέτρηση του οφθαλμού στα δίχτυα, τεχνικούς κανόνες για το νήμα που φτιάχνονται τα δίχτυα, όπως επίσης και ε, ποια είναι τα εξαρτήματα που μπορεί να επηρεάζουν ή να μειώνουν το άνοιγμα οφθαλμού, κατάλογο σκαφών που έχουν ε, την άδεια να φέρουν δοκότρατα και τεχνικοί κανόνες για την μέτρηση των εξαρτημάτων των εργαλείων αλίας και των, της μέτρησης των οφθαλμών και τα προσωρινά μέτρα διατήρησης αποθεμάτων ό, όταν χρειάζεται άμεση δράση. Ελπίζουμε αυτά να σας είναι σαφή και ίσως είναι κάπως τεχνικά, αλλά πιστεύουμε πώς θα καταφέρουμε να κλείσουμε αυτή την ε, πρόταση πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νικολέος που δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος βουλευτής που να θέλει κάτι να πει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τις προσπάθειες διευκρίνησης της Επιτροπής για να ε, εξηγήσει ποιες είναι ε, οι πράξεις και πράξεις εκτελεστικές και που αναφέρει ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις προκειμένου να γίνουν προπαρασκευαστικές εργασίες για τις οι πράξεις και αυτή η αιτιολογική σκέψη επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει νομίζω, <clears throat> να κατησυχάσουμε το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση αυτών των κατεξουδότητων πράξης και να φύγουμε από αυτή την δία ε, εμπλοκή που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα όμως ε, που αφορά το άρθρο 45. Εφόσον τελικά για αυτό το άρθρο βλέπουμε ότι για κατεπήγοντα μέτρα τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο ή μάλλον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δύο πράξεις, κατεξοδότηση ή κατεκτέλεση, και θα να θέσω το ερώτημα στην Επιτροπή για να μας πει πώς βλέπει την πραγματική εφαρμογή αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, χρειάζονται συνορματικά μέσα ε, τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους συμπληρωματικά. Αφού κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο, ας απαντήσει η Κομισιόν στα όσα Καταλάβαμε καλά το ερώτημα. Αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα εκδώσει κατεξοδόνση πράξης ή κατεκτέλεση. Οι πράξης πράξης προβλέπεται, χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν αλλαγές στα αποθέματα, αλλά δεν έχουν, έχουν άμεση εφαρμογή, αλλά δεν είναι απαραίτητο άμεσες. Όταν απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση, τότε προτείνουμε τις εκτελεστικές πράξεις. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Αν θέλετε, μπορούμε κατηδίαν να το συζητήσουμε αργότερα. Εντάξει. Ωραία, αφού δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, που είναι το σημείο 11, είναι η σύνδεση των υπερπόνιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης. Ξέρετε λοιπόν πως ο εισηγητής τον προηγούμενο μήνα συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα, να ενημερωθούμε και ο κύριος Ριβελίνη θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες και να σας πω πως για την κατάθεση τροπολογιών η προθεσμία λήγει 3 Ιανουαρίου το μεσημέρι. 3 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Ο κύριος Ριβελίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άρα το γεγονό 3 Ιανουαρίου το μεσημέρι είναι ακριβώ μετά τι γιορτέ. Αυτή η προθεσμία είναι κάπω παράδοξη, θα έλεγα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι υπερπώντε χώρε και εδάφη είναι ε, τα νησιά του Ατλαντικού, της Ανταρκτική, της Καραβική, του Ινδικού ωκεανού και του Ειρηνικού ωκεανού και εξαρτώνται συνταγματικά από τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δανία, τη Γαλλία, τις κάτω και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να αναδιατυπώσει τις αρχές από τι οποίε διέπεται η συνεργασία τη με τι ε, υπερπόντες χώρε και δάφη προσπαθώντας να προαγάγει την προσέγγιση και τις διτερότητε αυτών των χωρών. Στα πλαίσια τη ενωπημένη διαχείρισης των παρακτήων ζωνών, η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΙΧΕ ε, οδηγεί στην ανάληψη πολλών δραστηριοτήτων, οικονομικών, ε, αλληλευτικών, τουρισμού, μεταφορών και οι δυνατότητες που έχουν οι παράκτιες ζώνες όσον αφορά τις ΑΠΕ και τις πρώτες ύλες, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αναφορικά με τις θαλάσσιες υποθέσεις, η συνεργασία αυτή πρέπει να προάγει τη γνώση για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοτεχνολογία, την ενέργεια των ωκεανών, τη θαλάσσια επιτήρηση, τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και τη διαχείριση με βάση το οικοσύστημα. Όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των αλλιευτικών αποθεμάτων, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερπών χωρών και εδαφών πρέπει να βασίζεται σε μια υπεύθυνη διαχείριση τη αλληλεία στον τομέα τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των ελληνικών πόρων με τακτικέ διαβουλεύσει μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να γίνεται σωστή διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πόρων. Ω προ το τομέα τη αλίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει περισσότερο τα τοπικά συστήματα ελέγχου, επιτήρησης και επίβλεψή για να καταπολεμήσει την παράνομη αλία, την μη δηλωμένη και, φυσικά ε, το παράνομο εμπόριο που απορρέει. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία με τις περιφερειακές οργανώσεις ε, που διαχειρίζονται την αλία για να προωθηθούν μέτρα καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλίας που αυτή τη στιγμή αποτελούν μία από τις πιο μεγάλες απειλές για την βιωσιμότητα των πόρων και της βιοπικιλότητας ε, ε, της αλίας για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και των υπερπόντιων εδαφών και για να αντιμετωπιστεί αυτή η παράνομη αλία, έχω υποβάλει μια τροπολογία που αλλάζει το άρθρο 19.2 β της πρότασης της Επιτροπής και παρακαλώ τους συναδέλφους να διαβάσουν καλά το περιεχόμενο και να εγκρίνουν την τροπολογία ενδεχομένω. Ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο κάποιος όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, δεν θέλετε το λόγο. Τους έπεισα όλους, λέει ο κ. Όλα είναι ξεκάθαρα, λέει ο πρόεδρο. Όσον αφορά τώρα την προθυμία και τι τροπολογίε, κ. Βελίνη, το πρόβλημα είναι ότι η ψήφιση αυτή την Επιτροπή προβλέπεται για τι 21 Ιανουαρίου που θα συνεδριάσει η Επιτροπή μα. Γιατί στην ΤΕΒΕ θα ψηφίσουν τον Φεβρουάριο, οπότε μπορεί να μην έχουμε χρόνο να το κάνουμε πριν την συνεδρίαση της, ε, της 9 του Φεβρουαρίου. Άρα για να μπορέσουμε να, το, να στείλουμε, το, το, το, το, το Μάρτιο στην Ολομέλεια. <coughs> Οπότε δεν έχουμε στα διάφορα κάτι. Αν έχετε κάτι για τα διάφορα, τίποτε. Α, η κυρία Φράγκα. Όχι. 13 ανακοινώσει του Πρόεδρου για τι αποφάσει των συντονιστών. Κυρία Φράγκα, χωρί μικρόφωνο. Συζητήσαμε και είπαμε να εγκριθεί ένα σχέδιο προγράμματο για την ε, ε, ακρόαση όσον αφορά τα βαθύδια είδη. Γιατί αυτή η πρόταση δεν είναι τόσο καλά σταθμισμένη. Και ας πούμε σε ένα σήμα λέει ότι ακριβώς το πιο σημαντικό πρόγραμμα το οποίο το η Κομισιόν είναι ακριβώς το πρόγραμμα που ασχολείται με αυτά τα, ψάρια. Όμως εδώ αναφέρει το Ερμιόνι. Δεν έχω τίποτα κατά του Ερμιόνι. Αλλά είναι λιγότερο ενδιαφέρον από τα άλλα. Γιατί το, το πρόγραμμα, το πιο σημαντικό, δεν, δεν περιέχεται εδώ. Αυτό το Deep Fish Man που είναι αυτό το πρόγραμμα για αυτού του τα ψάρια. Άρα θα πρέπει να θίξουμε αυτό το πρόγραμμα, να ασχοληθούμε με αυτό, το οποίο ε, είναι, είναι το, το πιο κομικό σε αυτή την περιοχή. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κριτήριο για να μπορέσουμε να κάνουμε την αξιολόγηση. Δεν θέλω να επικρίνω αυτά που ήδη καλύπτονται, αλλά θα πρέπει να καλυφθούν και άλλα, να είναι επομένω πιο εξισορροπημένη η αντιμετώπιση. Το Deep Fish Man είναι το πιο μεγάλο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης αυτό αφορά και το άλλο πρόγραμμα, το Νηρέας, κάπως έτσι, το οποίο ακριβώς και λύσει τη χαρτογράφηση της περιοχής. Εγώ, ηλεκτροτρομά, θέλω να έρθω να συμφωνήσω με την κυρία Φράγα. Κυρία Λόβιν θέλω να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα το ξέρουμε. Εδώ και δύο εβδομάδες εγκρίθηκε από τους συντονιστές και το ξέραν και δύο συντονιστές της ομάδας σας. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες, οι σύμβουλοι συνεδρίασαν και όλοι είναι υπέρ. Άρα γιατί τώρα να αλλάξουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Πρόεδρος. Δεν είπε κανείς ότι δεν τήρηθηκε η διαδικασία. Ναι, έγιναν οι συναντήσεις που οι προτάσεις των πολιτικών ομάδων είχαμε 7 προτάσεις, μείνανε 6 κλπ. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Φράγα είναι το εξή. Χωρίς να θίξουμε τα υπάρχοντα, να το διευρύνουμε. Να βάλουμε άλλα δύο προγράμματα. Και να είναι πιο πλουραλιστική η πρόταση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Η μόνη αμφισβήτηση, η μόνη αμφιβολία που διατηρώ είναι ότι Δεν ξέρω αν θα κοστίσει, δεν θα κοστίσει το να προσθέτω τα δύο προγράμματα. Αλλιώ καμία αντίρρηση. Δεν θα βγάλουμε δύο για να βάλουμε άλλα δύο. Θα αυξήσουμε τα καλυπτόμενα. Αυτό ήταν η πρόταση. Υπάρχει πρόβλημα τεχνικό. Κύριε Λόβιν. Δεν είναι ορθό διαδικαστικά να λάβουμε τέτοια απόφαση εδώ και τώρα μια που είμαστε μόνο έξι. Το αποφάσισαν αυτό όλοι οι συντονιστές. Ήτανε όλοι εκεί. Γιατί τώρα να το αλλάξουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, οι αποφάσεις των συντονιστών κρίνονται εδώ στο σύνολό τους από τα μέλη της Επιτροπής. Είτε είναι εδώ, είτε δεν είναι. Και αυτοί που λείπουν είναι πρόβλημά τους. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Δυστυχώς είμαστε μόνο Έξι. Και δεν είναι αυτό και τόσο σπανία. Αυτό <clears throat> σίγουρα είναι ντροπή για τον πρόεδρο, σε οποιοδήποτε πρόεδρο. Οπότε, επαναλαμβάνω, οι αποφάσει των συντονιστών αν, ε, αναπέμπονται κατά κάποιο τρόπο στην Επιτροπή και η οποία κρίνει από τα μέλη της Επιτροπής, από αυτούς που είναι και όποιοι δεν είναι, δεν είναι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να έρθει να μην έρθει. Γι' αυτό σας λέω είχαμε αυτή την πρόταση και φυσικά μπορούμε να τη θέσουμε σε ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα που μάλλον δεν υπάρχει, είναι μια πρόταση διεύρυνσης της πρότασης κατά δύο προγράμματα επιπλέον. Αφέρετε το λόγο κύριε. Συγγνώμη πρόεδρε, αλλά δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά της κυρίας Φράγκα. Αλλά τώρα Τώρα το πήραμε το έγγραφο. Δεν ξέρουμε ε, περί τίνο πρόκειται καλά. Έχει γίνει αυτή η πρόταση να προσθεθούν άλλα δύο. Και αυτό θέλετε να ψηφίσουμε. Ναι, ναι, αυτό, αυτό λέει ο Πρόεδρος. Ε, εντάξει, άλλα δύο. Χωρίς να θίξουμε, λέει ο Πρόεδρος, αυτά που προβλέπονται και εγκρίθηκαν. Άλλοι δύο και άλλα δύο. Ποιοι συμφωνούν. Κατά αποχές άρα εγκρίνεται η πρόταση και επομένως θα προσθεθούν αυτοί οι δύο που προτάθηκε. Κάτι άλλο σε σχέση με τις αποφάσεις των συντονιστών. Τίποτε. Πολύ ωραία. Επομένως τώρα. Εντάξει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. αλλά η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 21 Ιανουαρίου και στις 22. Αυτά. Επομένως σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλές διακοπές, καλές γιορτές και να έρθετε ξανά εδώ ανανεωμένοι και με ενέργεια του χρόνου. Κάθε ευχή σε όλους. Για όλους, θα λέω για όλους ενώ Όλους που εδώ και τους διερμηνείς.